Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. So, it's our pleasure this afternoon to uh, Με μεγάλη χαρά, σήμερα το απόγευμα θα καλωσορίσουμε τον Επίτροπο κύριο Βέλα, θα κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων και έχω και μία παρατήρηση για τα πρακτικά θέματα πριν ακούσουμε τον Επίτροπο, στις 4 θα ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν μην ξεχάσετε, χρειάζεστε την κάρτα για τις ψηφοφορίες, γιατί μόλις τελειώσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο θα περάσουμε στην ψηφοφορία και όποιος δεν έχει την κάρτα του δίπλα του θα δυσκολευτεί, δεν θα προλαβαίνει. Οπότε ζητήστε από τους συναδέλφους σας ή από ε, τους βοηθούς σας να σας φέρουν τις κάρτες να είναι έτοιμες. Επανέρχομαι λοιπόν, σας καλωσορίζω, χαίρομαι πάρα πολύ που θα είστε εδώ, που θα σας ακούσουμε, που θα ακούσουμε και το ποιες είναι οι προτεραιότητες των δικών μας μελών για την βιοπικιλότητα. Τα όσα έκαναν ε, και έγιναν φέτος το καλοκαίρι επανέφεραν την βιοπικιλομορφία σε, ε, στην επικαιρότητα και είναι προφανές ότι μέχρι την κόπ της Κίνας το 2020 η βιοπικιλότητα θα το συζητάμε το θέμα όλο και περισσότερο και ξέρετε πως το ίδιο έγινε και με το κλίμα πριν από μία δεκαετία μετά τη συνάντηση ε, είχε μεγαλύτερη ορατότητα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα συζητάμε περισσότερο τη βιοποικιλότητα και λιγότερο το κλίμα, γιατί στο κλίμα όλοι αισθανόμαστε ότι κάποιε κινήσει γίνονται και υπάρχει και ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, που είναι κομβικό, γιατί το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και στο εσωτερικό θεματολόγιο αλλά και στο εξωτερικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ λοιπόν που είστε εδώ, που θα σας ακούσουμε Ξέρουμε πως δεν μπορείτε να αναλάβετε νέες υποχρεώσεις για την επόμενη θητεία, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μία απογραφή μετά το πέρας της θητείας σας, για να ε, ενημερώσουμε και τα νέα μέλη της Επιτροπής μας και να τους δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το υπόβαθρο. Σας ευχαριστώ πολύ. 10-15 λεπτά και μετά θα κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, Πασκάλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι χαρά για μένα να έρχομαι σε αυτή την επιτροπή σας με τη νέα σύνδεση, να συγχαρώ όσους είναι καινούργοι και να καλωσορίσω τα παλιά μέλη με τα οποία είχα τη χαρά να συνεργαστώ τα τελευταία πέντε χρόνια. Ξέρω πως ενδιαφέρεστε πολύ για τα θέματα του περιβάλλοντος και γνωρίζω πως ενδιαφέρεστε για την αυριανή συζήτηση με τα ε, μέλη του προσωπικού της δικής μου Γενικής Διεύθυνσης για θέματα ε, περιβάλλοντος. Σήμερα ε, μιλήσατε για τα χημικά. Έχετε αύριο να θέσετε το θέμα της αποψήλωσης και των περιβαλλοντικών μέτρων. Οπότε έχω δώσει οδηγίες να σας ενημερώσουν για όλα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ρωτά τι κάνουμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Οι πολίτες μας και πιο πολύ η νέα γενιά ζητάνε από μας που χαράσουμε πολιτικοί να είμαστε πιο αποφασιστικοί όταν αντιμετωπίζουμε τα θέματα του περιβάλλοντος. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό αποκτάτε περισσότερη στήριξη από το εκλογικό σας σώμα, αλλά ε, είστε και όλο πιο υπεύθυνοι. Όταν ξεκίνησα την παρουσίασή μου ε, πριν από πέντε χρόνια, είπα ότι δεν κληρονομούμε το περιβάλλον και τον πλανήτη από τους γονείς μας, αλλά το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας. Και θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να τους αφήσουμε ε, ένα καλύτερο πλανήτη και στα παιδιά μας ε, και στα εγγόνια μας. Αντιμετωπίζουμε δύο μεγάλες προκλήσεις για το πολιτισμό μας και την ανθρωπότητα. Απόλυα βιοπικιλότητας και αλλαγή του κλίματος. Η απώλεια αυτή τη στιγμή βιοπικιλότητας είναι η μεγαλύτερη ε, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Πάνω από ένα δις ήδη μπορεί να εξαφανιστούν λόγω ε, μη βιώσιμης ανθρώπινης ε, δραστηριότητας. Είναι μαζικές αυτές οι καταστροφές. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάτι ανάλογα στο παρελθόν και μπορεί να μην είναι ε, αναστρέψιμο. Από τη μελέτη που έχω πει και τα στοιχεία της IPB, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αν δεν ε, κάνουμε μια ριζική ε, αναστροφή αυτής της απώλειας, οι στόχοι που έχουμε βάλει για τη βιωσιμότητα είναι αδύνατο να επιτευχθούν. Άρα λοιπόν το θέμα επήγε. Ο χρόνος πιέζει. Η αξιολόγηση που έγινε από την IBB επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα για απώλεια φυσικού περιβάλλοντος με έναν ρυθμό άγνωστο στο παρελθόν. Οι φωτιές στα δάση του Αμοζονίου... μας δείχνουν ποια είναι η πραγματικότητα για την αλλαγή την περιβαλλοντολογική, όπως επίσης και την απώλεια βιοπικιλότητας. Αυτή τη στιγμή μας ζητάνε όλο και περισσότερο να αναβάλουμε δράση. Ε, στο Ευρωβαρόμετρο ε, φάνηκε πως μία από τις πέντε βασικές ανησυχίες των πολιτών στην Ευρώπη είναι το περιβάλλον, πάνω ακόμα και από την ανεργία. Θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε με τόλμη αυτές τις ε, τεράστιες αλλαγές με μέτρα που θα καλύπτουν όλο το φάσμα ε, πολιτικών. Τώρα το βασικό όχημα δεν έχει αλλάξει, αλλά παρόλες τις ε, δράσεις μας δεν έχουμε κάνει κάτι το οποίο είναι αρκετό για να αναστρέψει αυτή την ε, χειροτέρευση ε, της βιοπικιλότητας. Ίσως γιατί δεν έχει ενταχθεί σε όλες τις βασικές πολιτικές. Εμείς θα πρέπει να ηγηθούμε μέσω του παραδείγματος που θα δώσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί αν θέλουμε να κάνουμε κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να τους δείξουμε τι πετυχαίνουν τα δικά μας εσωτερικά μέσα οδηγίες οι σχετικές αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο αυτής της πολιτικής. Και αν θυμόσαστε καλά, όταν ξεκίνησα πριν από πέντε χρόνια την εντολή μου, ε, ανέλαβα να κάνω μία εισεβάθος αξιολόγηση αυτών των οδηγιών. Τα ευρήματα από αυτή από αυτόν τον έλεγχο καταλληλότητας είναι ε, σαφές το νομικό πλαίσιο είναι ε, σταθερό. Και σε συμφωνία με ε, τον συνομοθέτη και την κοινή γνώμη δεν προτείναμε να ε, τροποποιηθούν. Παρ' αυτά έχουμε μεγάλα προβλήματα με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των οδηγιών. Και παρόλο που σε κάποιες περιοχές και οικοσυστήματα πολύ πλούσια της Ευρώπης προσφέρουν βασική στήριξη, δεν καλύπτουν όλες τις άλλες γωνιές της Ευρώπης πέραν των οικοσυστημάτων ε, Natura. Προσπαθήσαμε μέσω του σχέδιου δράσης για ε, τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία να δώσουμε κάποιες λύσεις. Και κάποιοι στις χώρες τους δημιούργησαν μακροπρόθεσμα ε, πλαίσια για να εντάξουν τις περί ε, φύσης ε, οδηγίες και να προστατεύσουν το περιβάλλον. Χτες παρουσιάσαμε ε, τις αναμενόμενες κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε πώς μπορούμε στις διάφορες αποφάσεις να εντάξουμε τα θέματα αυτά. Το να κλείσουμε το δίκτυο Natura 2000 και σε επίπεδο χερσαίο και θαλάσσιο είναι ο βασικός μας στόχος. Για τα θέματα αυτά έχουμε προχωρήσει πολύ τα τελευταία πέντε χρόνια και πρέπει να σας πω όχι μόνο στο να εντοπίσουμε ποιες είναι οι περιοχές Natura, αλλά στο πώς να τις διαχειριστούμε. Και να σας πω πως το ποσοστό των ε, εκτάσεων που προστατεύονται έχει ανέβει από το 50% στο 70% που είναι υψηλό. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να βελτιωθούν. Και γι' αυτό έχουμε κάνει προσπάθειες επιβολής. 17 διαδικασίες επί παραβάση, πάνω από 30 έρευνες. Αυτά τρέχουν σήμερα έτσι ώστε να πιέζουμε και να εξασφαλίζουμε πως τους κανόνες θα τους εφαρμόζουν σωστά. Επίσης θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους για να έχουμε μεγαλύτερη συμμόρφωση και μέσω ε, διαλόγου για να έχουμε αρκετές επενδύσεις, αυτό που είναι απαραίτητο είναι να εξασφαλίσουμε πως τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι διαθέσιμα. Και εδώ ο δικός σας ρόλος είναι κρίσιμος και πιο συγκεκριμένα για τις ε, διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για την ΚΑΠ. Το αποτέλεσμα θα ε, διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό την υγεία του περιβάλλοντος ε, στην Ευρώπη γιατί ο τρόπος χρήσης γης στη βιβλιοκαιλότητα και στην απώλεια αυτής είναι ε, από τα πιο βασικά σημεία. Για την Γεωργία θα τα πω με μεγαλύτερες λεπτομέρειες αργότερα. Να πω κάτι όμως και για τους ωκεανούς και τις θάλασσές μας. Μετά τη δημοσίευση της στρατηγικής ε, για ε, τη θάλασσα και τις σχετικές οδηγίες και πιο συγκεκριμένα όλα τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε κάνει πολλά για να προστατεύσουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Παρόλα αυτά το θαλάσσιο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζει ανησυχητικά φαινόμενα χειροτέρευση και το να φτάσουμε σε μια καλή κατάσταση μέχρι το 2020 για όλα τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θαλάσσια, δεν μοιάζει να είναι ε, εύκολο να επιτευχθεί. Ε, χάρη στις, ευκαιρί... στις ε, προσπάθειες που έγιναν για να εφαρμοστούν οι κανόνες μας και να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον, σχεδόν διπλασιάσαμε ε, τις θάλασσές μας που θεωρούνται προστατευόμενος θαλάσσιος χώρος. Δηλαδή από το 6% πριν από 7 χρόνια φτάσαμε στο περίπου 11% σήμερα. Ξεπερνώντας λοιπόν το στόχο που ήταν το 10%. Όμως έχουμε μεγάλες περιφερειακές διαφοροποιήσει και χρειάζονται παραπάνω προσπάθειες. Τα απόβλητα στη θάλασσα. Τεράστιο πρόβλημα για την θαλάσσια βιοποικιλότητα και για την υγεία των ωκεανών μας. Η οδηγία για τα πλαστικά μιας χρήσης ε, που πέρασε σε χρόνο ρεκόρ στα πλαίσια της στρατηγικής για τα πλαστικά είναι το πιο σφαιρικό νομικό εργαλείο παγκοσμίω που λύνει το θέμα των αποβλήτων, των πλαστικών αποβλήτων στη θάλασσα. Έχουμε όμως και τα μικροπλαστικά και εκεί πρέπει να κάνουμε κάτι για να είναι υγιείς οι ωκεανοί. Τι έχω κατά νου. Μιλάμε για τα πλαστικά που πετάνε ε, ε, στις, θάλασσες, αλλά δεν μιλάμε καθόλου ε, για ε, ε, κάποια στοιχεία, ηχνοστοιχεία τα οποία πετάμε στις θάλασσες, που είναι πολύ πιο βλαβερά. Να δούμε τώρα και το θέμα της ΚΑΠ. Ο ρόλος της ΚΑΠ είναι να αντιμετωπίζει και τα οικονομικά και τα περιβαντολογικά προβλήματα της βιωσιμότητας υγειοργίας. Οι προτάσεις για την ΚΑΠ 21-27 από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθεί να θέσει την ε, περιβαλλοντολογική προστασία στην καρδιά τη στρατηγική της για να λύσουμε το, και για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ε, με το κλίμα και την βιοποικιλότητα και να έχουμε μια πιο βιώσιμη γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω λοιπόν κάποια στοιχεία. Οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις άμεσες επιδοτήσεις η ερεσιμότητα δηλαδή έχει ενισχυθεί, όπως επίσης και τα θέματα βιοπικιλότητας. Οπότε ε, ε, ε, για τις μόνιμους βοσκότοπους και για τις βαλτόδες περιοχές ενισχύεται στα πλαίσια της Natura 2000 η προστασία. Επίσης, άμυψης φορά και σχετικές υποχρεώσεις. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως οι επιδοτούμενοι γεωργοί στην Ευρώπη συνεισφέρουν στην προστασία της βιοπικιλότητας. Δεν μπορούμε να δίνουμε εξαιρέσεις. Η χειροτέρευση στην βιοπικιλότητα θα πρέπει να αναστραφεί και θα το λάβουμε αυτό υπόψη γιατί έτσι θα γίνει μακροπρόθεσμα βιώσιμη η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερα κίνητρα για φιλικέ προ το περιβάλλον προσεγγίσεις. Η μεγάλη καινοτομία στη νέα ΚΑΠ είναι τα οικολογικά καθεστώτα στον πρώτο πυλώνα. Eco schemes με άμεσε ενισχύσει που θα πληρώνονται στι εκμεταλλεύσει έτσι ώστε να στηρίζονται πρακτικέ που είναι προ όφελο τη βιοπικιλότητα. Τρία κομβικά στοιχεία στι προτάσει μα εξασφαλίζουν ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαντολογικής φιλοδοξίας. Πρώτα απ' όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει για το περιβάλλον και για το κλίμα να οριοθετήσουν, το, να περιχαράξουν το 30% των ε, ε, κονδυλίων που έχουμε στο δεύτερο τους πυλώνα για την, ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη. Στα στρατηγικά σχέδια για την ΚΑΠ χρειάζεται μεγαλύτερη συνεισφορά ε, έτσι ώστε να επιτύχουμε συγκεκριμένους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον. Και τέλος, θέλει μία αποτελεσματική εμπλοκή των ε, περιοντολογικών αρχών ε, στην ε, προετοιμασία των στρατηγικών σχεδίων, των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, έτσι ώστε να έχουμε συνέργειες για τις στρατηγικές βιοπικιλότητας, οι οποίες θα αναλαμβάνονται σε επίπεδο κράτους μέλους. Δεν χρειαζόμαστε μόνο περισσότερα κονδύλια για τη βιοπικιλότητα, χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματική δαπάνη αυτών που έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα, για την περιβαλλοντολογική αποτελεσματικότητα της ΚΑΠ, να σας πω ότι εξαρτάται καταρχήν από το σε ποιο βαθμό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα στηρίξουν τις περιβαλλοντολογικές φιλοδοξίες της νέας ΚΑΠ και δεύτερον από τις επιλογές που θα κάνουν τα κράτη-μέλη στα πλαίσια των εθνικών σχεδίων για την ΚΑΠ μια και η νέα ΚΑΠ έχει πολύ περισσότερα στοιχεία επικουρικότητας και, ε, και ε, έχουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη τα κράτη-μέλη. Σήμερα θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω μια έκκληση προς εσάς. Η φιλοδοξία ε, των διατάξεων για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ να παραμείνει και να μην μειώσετε ή διαγράψετε αυτά που προτείνουμε. Τι λέμε για τη στρατηγική για την ποικιλότητα για το 2020. Λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και της κρίσης στο περιβάλλον, το να συνεχίσουμε όπως το παρελθόν δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο από ε, κάποιες ε, μικρές βελτιώσεις. Η Ursula Βαντελάιν έχει υποσχεθεί πως θα είναι φιλόδοξο το Green Deal και η περιβαλλοντολογική της πολιτική και υποσχέθηκε να παρουσιάσει εν ώψη του 2030 μια νέα ε, στρατηγική για τη βιοπικιλότητα. Εγώ έχω ήδη απευθύνει έκκληση στα κράτη-μέλη σε ένα πρόσφατο συμβούλιο για το περιβάλλον για να συζητήσουν με άλλους βασικούς πολιτικούς κλάδους και να δούμε ποιο θα είναι το μέλλον της βιοπικιλότητας και αυτό θα έπρεπε να ισχύει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα πρέπει ε, αυτή την απώλεια να την αναστρέψουμε μέσω κάποιας τολμηρής αποτελεσματικής συνεισφοράς μέσω της γεωργίας, της εμπορίου, της βιομηχανίας αλλά και της οικονομικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα έφτασε πια η ώρα να δούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και όπως είπε ε, στις νέες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να έχουμε εγκάρσια πρότυπα τα οποία να ισχύουν για την βιοπικιλότητα. Όραμά μου θα ήταν να πετύχουμε αυτούς τους στόχους με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιευσήψαμε χτες, με μια ολοκλήρωση των συστημάτων, ε, των, ε, της διαχείρισης οικοσυστημάτων μέσα σε ένα πιο στεναρό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να πλαισιώσει τις υφιστάμενες ε, οδηγίες για την φύση και να έχουμε μια πιο διευρυμένη ε, πλειάδα μέτρων που θα μας επιτρέπει ε, να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη και να αναστρέψουμε ε, την απώλεια βιοποικιλότητας. Δηλαδή, ένα μέλλον για τη βιομηχανία και για το περιβάλλον που θα έχει συστήματα λογοδοσίας και σε επίπεδο που θα λαμβάνουν υπόψη και το φυσικό μας κεφάλαιο έτσι ώστε να έχουμε βιώσιμη χρηματοδότηση, έτσι ώστε και εμείς να βγούμε ε, στην επίθεση ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, εμείς θα μπορέσουμε να αποδείξουμε πόσο στρατευμένοι είμαστε υπέρ του περιβάλλοντος στην COP15 ε, τον Οκτώβριο του 2020 στην Κίνα, όταν η μετά το 2020 προσέγγιση για την βιοποικιλότητα εγκριθεί τους ε, στόχους του 2010 τους χάσαμε. Θα χάσουμε και τους στόχους του 2020. Δεν μπορούμε να ξανααποτύχουμε αργότερα. Θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να λέει λιγότερα και να κάνει περισσότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η νέα υποεκλογή πρόεδρος θα πρέπει με τους παγκόσμιους εταίρους μας να προσπαθήσει τα επόμενα πέντε χρόνια να περιορίσει την απώλεια βιοποικιλότητας και να επιτρέψει η COP για ε, του 2015 να είναι εξίσου επιτυχής με την COP για τη διάσκεψη για το κλίμα για το, στο Παρίσι. Να είναι μια φιλόδοξη στιγμή με στόχους οι οποίοι θα είναι μετρήσιμοι, φιλόδοξοι, θα είναι δεσμευτικοί ε, για τους εταίρους και με ένα μηχανισμό ενδιάμεσης αναθεώρησης με πυγμή βασικός μας στόχος παρόμοιος με αυτά τα οποία βάλαμε για την αλλαγή του κλίματος και με στήριξη πολιτική. Παρόλο που η επιστημονική συζήτηση είναι περίπλοκη, πιστεύω πως ο στόχος είναι απλός. Ένα εκατομμύριο ε, που εξαφανίζονται είναι ένα εκατομμύριο παραπάνω ήδη από αυτά που θα έπρεπε να εξαφανίζονται. Και είναι ένα θέμα στο οποίο θα μας στηρίξουν οι πολίτες, όλου του πλανήτη. Η βιοπικιλότητα χρειάζεται να ε, προστατευτεί και ε, στις ε, χερσαίες περιοχές αλλά και στις θαλάσσιες και γι' αυτό στο θεματολόγιο της διαχείρισης των ωκεανών χρειαζόμαστε, όπως έχω πει, μια νέα συμφωνία που θα προστατεύει και στην ανοιχτή θάλασσα τη βιοπικιλότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήταν τόσο θετικό το αποτέλεσμα των συζητήσεων στις τελευταίες διαπραγματεύσεις που έγιναν για τη συμφωνία αυτή που, έκλεισα που τελείωσαν την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Παρ' όλα αυτά, μακρύς ο δρόμος, έτσι ώστε να έχουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι εύχριστη και φιλόδοξη. Να σας πω όμως πως για το μέλλον θέλω να επανέλθω σε μια πολύ ανησυχητική απειλή που είναι οι συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Αμαζονίου και όχι μόνο εκεί. Είχαμε και στην περιοχή του Αρκτικής και στη Σιβηρία και στην Ελλάδα και στην Αφρική. Αυτές οι πυρκαγιές μας υπενθυμίζουν πόσο έθραυστα είναι τα δασικά οικοσυστήματα και είναι δική μας ευθύνη να τα προστατεύσουμε. Είναι απαραίτητα τα δάση, όχι μόνο για να στηρίξουμε τους νόμους, αλλά γιατί αποτελούν ε, απαραίτητο συστατικό των ανθρώπων που ζουν ε, στην Ήπεθρο. Ε, και είναι η βασική τους οικονομική δραστηριότητα. Και ξέρετε πως η αποψήλωση των ε, ε, δασών είναι ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την αλλαγή του κλίματος μετά τα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε μείνει πίσω. 800 γήπεδα ποδοσφαίρου χάνονται κάθε ώρα τα τελευταία 30 χρόνια. Η γεωργική επέκταση είναι το 80% της ε, παγκόσμιας ε, αποψήλωσης δασών. Και το και εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνουμε το 1 τρίτο των γεωργικών προϊόντων και άλλων προϊόντων που παράγονται από αυτές τις από, ε, ψηλωμένες γέες. Άρα λοιπόν είμαστε ε, και η Ευθύνη, αλλά θα πρέπει να έχουμε και πολλά προγράμματα δάσωσης για να το αναστρέψουμε αυτό. Έχει ξεκινήσει η ευρωπαϊκή δράση ε, και έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ε, ξαναζήσουν τα παγκόσμια δάση. Την παρουσιάσαμε στην αρχή του καλοκαιριού και ζήτησα από τη συνάδελφο Άστριντ από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος να σας ενημερώσει πιο συγκεκριμένα ε, θέματα αύριο. Ξέρω πως θέλατε να σας πω ε, και δύο για τη σύμβαση sites, να σας πω κάποια βασικά αποτελέσματα, ε, αλλά μπορούμε να τα πούμε και αργότερα. COP18, σύμβαση sites, έκλεισε στη Γενέβη την περασμένη εβδομάδα και είμαι ικανοποιημένο από τα αποτελέσματα. Ήταν η συνάντηση των συμβαλωμένων μερών. Παίξαμε πολύ σημαντικό ρόλο. Κανένα μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν στην αντιπροσωπεία μα αυτή τη φορά. Γνωρίζω όμω πω αρκετοί από εσά παρακολούθησαν τη διάσκεψη αυτή στενά. Όλε οι προτάσεις μας για επιπλέον ήδη ε, στη σύμβαση εγκρίθηκαν και τις περισσότερες φορές ομόφωνα. η διάσκεψη εισήγαγε ε, εμπορικούς περιορισμούς για το εμπόριο ε, ζωικών και φυτικών ειδών, για παράδειγμα κάπιλοπαρδάλης, αλλά και καρχαρίες, ε, θαλάσσια αγκούρια ή καλκάνια. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα προστατεύσουμε γιατί αν λαμβάνουμε υπόψη τους στόχους αυτού σοβαρά, το εμπόριο των ειδών αυτών θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά. Επίσης, συνεργασία με, άλλους, με άλλα συμβαλόμενα μέρη στην συμφωνία αυτή βοήθησε στο να πάμε καλά έχουμε ε, ρυθμίσει ε, την μεταφορά ε, των ελεφάντων της Αφρικής εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος και εδώ παίξαμε πολύ σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεση σε μια συμφωνία που προστατεύει τους ελέφαντες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς παρόλο και εξασφαλίσαμε πως ε, οποιαδήποτε τέτοια μετακίνηση ε, θα γίνεται σύμφωνα με ε, επιστημονικά κριτήρια όπου υπάρχει θέμα ευζοίας των ζώων και προστασίας του περιβάλλοντος. Θα ήθελα και στο μέλλον να συνεχίσουμε με αυτή την σφαιρική προσέγγιση έτσι ώστε να καθορίζονται οι κανόνες του εμπορίου για τα ζώα, για τα μεγάλα θυράματα πιστεύω πως θα πρέπει να το κάνουμε είτε σε πολυμερές είτε σε διμερές επίπεδο, δηλαδή και μέσω συμφωνιών όπως οι sites. Θα πρέπει οι διάφορες πολιτικές να μην έχουν στεγανά μεταξύ τους και ελπίζω πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να μας στηρίζει. Ευχαριστώ πολύ για να κλείσουμε σε όλα τα θέματα τα οποία ανέφερα. Βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στο δυναμισμό σας και στην ιδιαίτερη στήριξη εσάς που είστε μέλη αυτής της τόσο σημαντικής επιτροπής στα φιλόδοξα σχέδια που έχουμε. Ευχαριστώ. Άρα μας ζητάτε υποστήριξη και κίνητρα. Και ελπίζω και τα, τα μέλη μας, οι βουλευτές μας να σας προσφέρουν την υποστήριξη αυτή. Έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων. Συντονιστές των ομάδων. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ανιά Σεβά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την παρουσία σας και την παρουσία σας εδώ. Μας μιλήσατε για την ενίσχυση της προστασίας των ε, ελεφάντων της Αφρικής και νέων ε, ειδών που αποτελεί ένα θετικό βήμα με την ε, Σύμβαση για την Προστασία της Βιοποικιλότητας. Ωστόσο δεν πρέπει να σταματήσουν εδώ ε, στις ιτές δηλαδή και τη ρύθμιση του διεθνού συμπορίου αυτές οι προσπάθειες γιατί αποτελούν μόνο ένα πρώτο βήμα. Πρέπει να καταπολεμήσουμε και την, το λαθρεμπόριο άγριων ειδών που αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία των ειδών. 40.000 ελέφαντες ε, φωνεύονται κάθε χρόνο λόγω αυτού του λαθρεμπορίου και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε σημεία μετάβασης και διακίνησης των προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ως εκ τούτου έχει σημαντική ευθύνη στον τομέα αυτό. Κύριε Επίτροπε, το σχεδίο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ε, εκπνέει του χρόνου. Η έκθεση για, τις, ε, ε, για τα επιτεύγματα υπογραμμίζει πω πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών για να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020. Ερωτώ λοιπόν πολύ σύντομα αν μπορείτε να μα βεβαιώσετε πω θα υπάρξουν νέα μέτρα ή αν έχουν αναλυφθεί ήδη ενδεχομένω για να, καλυφθούν, να καλυφθεί το χαμένο έδαφο. Οι δέσιτε που συχνά χάνεται η αποτελεσματικότητά της σε κάποια κενά ή παραθυράκια από τα οποία μπορούν και κινούνται οι λαθροδιακινητές και εάν υπάρχει τρόπος να επιταχυνθεί η εναρμόνιση των κανονών μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που τηρήσατε το χρονικό όριο των δύο λεπτών. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Κυρία Γκούτλαντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Βέλα, που ήρθατε σήμερα και έτσι μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για το μέλλον και δει το πώς μπορούμε να αποτρέψουμε και να αναλάβουμε δράση όταν βλέπουμε αυτές τις καταστροφικές εξελίξεις στον τομέα της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Βρισκόμαστε σε μια εν εξελίξει οικολογική καταστροφή. Είναι σαφείς οι εκθέσεις που μας λένε ότι τα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο υφίστανται φοβερές πιέσεις. Είναι υποκατάρρευση. Η έκθεση της IBS είναι μια ακόμη στη σειρά πολλών τέτοιων μαρτυριών και βεβαίως ξέρω ότι είστε ενημερό και παρακολουθείτε τις εκθέσεις αυτές. Ωστόσο επισημαίνω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθυστερήσει ιδιαίτερα και δεν έχει κάνει ό,τι μπορούσε για την προστασία της βιοπικιλότητας. Ε, εξακολουθούμε να μολύνουμε το περιβάλλον μας με ζυζανιοκτόμνα, πλαστικά αλλά και άλλα προϊόντα που καταστρέφουν τη βιοπικιλότητα. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, πότε εσείς και η Επιτροπή θα καταθέσετε πρόταση για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες. Και γιατί η χρήση των ζυζανιοκτώνων δεν έχει περιοριστεί από τη δεκαετία του 90 παρά το γεγονός ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία προσδιορίζει στόχους και λειτουργία ε, μιας στρατηγικής. Επίσης μιλάτε για μικροπλαστικά. Βλέπουμε όμως ότι τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να αναλαμβάνουν ε, δράση. Επειδή υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, βλέπουμε νομοθεσία για τα καλλιντικά, τις οδοντόκρεμες. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας προστατέψει από τα προβλήματα αυτά που διαπιστώνουμε στο περιβάλλον λόγω των μικροπλαστικών. Η ΚΟΠ της Κίνας του χρόνου θα αποτελέσει ένα σημείο καμπής για ανάληψη διεθνών υποχρεώσεων υπέρ τη βιοπικιλότητα και σα αναφερθήκατε στα δάση πολύ ωραία. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα παρακολουθείτε διαλύπτω, ωστόσο. ερωτώ τι μπορούμε ακόμα να κάνουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει για ακόμα περισσότερη συγκεκριμένη αλλά και παγκόσμια δράση για την προστασία τη βιοπικιλότητα στην Ιφίλιο. Συμφωνείτε πως θα πρέπει η Ευρώπη να αξιοποιήσει κάθε δυνατή επιλογή και εμπορικέ συμφωνίες δηλαδή, ώστε και οι λοιποί παράγοντες ε, σε διεθνές επίπεδο χώρες και ε, ενός κρατών να αναλάβουν αντίστοιχη δράση και δεσμεύσεις. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ κύριε Βέλα που είστε εδώ, κύριο Στόρβαλτς. Πρόκειται μάλλον για μια από τις τελευταίες ευκαιρίες που έχουμε να συζητήσουμε μαζί. Ξεκινώντας λοιπόν με την καύση ορυκτών καυσίμων, παράγουμε περί τους 10 γιγατόνους το χρόνο. 150 γιγατόνι διοξιδίου του άνθρακα πάντα. Προέρχονται από τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο και αν κάτι πάει πράγματι στραβά είναι αυτό. Δεν θα μπορέσουμε να, το, να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. 25% της βιοπικιλότητας του κόσμου της Φιλίου βρίσκεται στην περιοχή αυτή του Αμαζονίου. Εμείς στη Φιλανδία έχουμε μια πολύ καθαρή φύση με τα αρκτικά δάση και μπορούμε να μιλούμε για βιοπικιλότητα αρκτικών δασών σε όρους μιλιγκράμμ, ε, χιλιοστογραμμαρίων ε, μάλλον, στην, ε, σε επίπεδο εκπομπών. Είχαμε μάλιστα ένα μορατόριο στη χρήση της σόγιας από το 2009 και αν κοιτάξει κανείς τα ποσοστά της, α, της δασών, της αποψηλούς δασών, βλέπουμε ότι και η συμφωνία και το μορατόριο έφεραν αποτελέσματα. Το, η αποψήλωση στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας, όσο τηρήθηκε αυτή η συμφωνία με το μορατόριο, έφερε α, ικανοποιητικά αποτελέσματα, μειώθηκε δηλαδή η αποψήλωση όταν ε, κάποιες κυβερνήσεις δεν κάνουν αυτό το οποίο οφείλουν, που έχουν αναλάβει δέσμευση και ευθύνε. Ε, και αυτό δεν αναφέρεται μόνο στην ηγεσία, αλλά και στις αγορές. Κινέζοι έχουν ένα ποσοστό καταναλώσεις βόηου κρέατος ισοδύναμου με αυτό των ΗΠΑ σχετικά χαμηλό, αλλά, έχουν ένα, αλλά είναι 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι που όλο και περισσότερο κρέας βόλιο καταναλώνουν, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η αγορά αναγκαστικά θα προσαρμοστεί και θα οδηγήσει σε συνέπειες αντίστοιχε με αυτέ που βλέπουμε τώρα στη Βραζιλία. Τι θα κάνετε λοιπόν γι' αυτό. Η κυρία Τουσάν, πράσινη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, οι πυρκαγιές ε, που μένονται στην Αμαζονία έχουν καταστρέψει 470.000 εκτάρια. Έχουν καταστραφεί δάση μοναδικά στον κόσμο. Και αυτό τι ήταν, ότι ήμασταν απλώς άτυχοι. Όχι. Υπάρχουν ε, υπεύθυνοι. Ναι, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Ναι. Οι πολυάριθμες πυρκαγιές δεν οφείλονται στην ξηρασία, αλλά σε οικονομικά συμφέροντα που, θυσιάζονται, όπου θυσιάζουν, που στο βωμό του θυσιάζεται η φύση. Γίνονται πυρκαγιές δηλαδή, προξενούνται πυρκαγιές έτσι ώστε να μπορέσει η βιομηχανία τροφίμων αλλά και ε, της δασοπονίας να εξασφαλίσει εδάφη για τα οικονομικά της συμφέροντα. Δεν ισχύει αυτό που μπορούσα να ότι ο Αμαζόνιος ανήκει ε, στο, στη Βραζιλία αλλά σε ολόκληρη την υφήλη. Ο Τσίκο Μέντες, αγωνιστής ε, του περιβάλλοντος ε, που δολοφονήθηκε το 1988, είχε πει τι έλεγε στην αρχή αγωνίστηκα για να σώσω μερικούς πληθυσμούς αυτού Στη συνέχεια αγωνιζόμουν για να σώσω τα δάση του Αμαζονίου. Τώρα αγωνίζομαι για, ολόκληρη, για ολόκληρο τον πληθυσμό της γης. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε λοιπόν ή να αποστρέψουμε το βλέμμα. Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι είμαστε και εμείς ε, συνυπεύθυνοι στη Γουιάννα προκειμένου να κάνει εξόριξη χρυσού η Γαλλία. οτι ειμαστε και εμεί συνυπευθυνοι στη γουιαννα προκειμενου να κανει εξοριξη χρυσου η γαλλια κανει τα στραβά μάτια στις αποψηλώσεις των δασών και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και εκεί, όπως και στην περίπτωση Βρασιλίας κατά τον Μπορσονάνο, πότε θα αναγνωριστεί δικαίωμα στη φύση, δικαίωμα της, ε, στην ε, προστασία της υφηλίου, πότε θα μιλήσουμε για οικολογικά εγκλήματα, πότε θα προστατέψουμε τον πλανήτη μας, πώς ε, σκοπεύει να απαντήσει σε μια όχι μόνο καταστροφική οικολογική κρίση, αλλά και σε μια βαθύτατη προσβολή των δικαιωμάτων που έχουμε σε μια καθαρή φύση. κυρία Λίμερ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Ποιος δεν θα ήθελε να προστατεύσουμε τη φύση, το περιβάλλον και να έχουμε βιοπικιλότητα. Από ό,τι κατάλαβα από εσάς, εδώ βρίσκομαι, ότι θέλετε να κάνετε τα πάντα για να ε, αποτρέψουμε την ε, εξαφάνιση των ειδών λόγω της ε, ανθρώπινης δραστηριότητας. Εδώ συζητάμε πολλά προβλήματα τα οποία δεν θα είχαμε αν δεν είχαμε και την ευρωπαϊκή πολιτική. Σήμερα ακούσαμε ότι μέχρι το 2050 θέλουμε να πετύχουμε ουδετερότητα όσον αφορά τη χρήση καυσίμων τα, στις αερομεταφορές. Έχουμε όμως ακριβώς ε, καλλιέργεια βιοκαυσίμων, ε, τα οποία απαιτούν εδάφη, τα οποία ε, αποκτώνται με την αποψήλωση των τροπικών δασών. Και αυτό δεν αφορά μόνο το φινικέλαιο, αφορά όλα τα βιοκαύσιμα που χρειάζονται τεράστιες εκτάσεις για την παραγωγή ενέργειας. Ή ας κοιτάξουμε και την Ευρώπη ακόμα. Ε, ολικές εγκαταστάσεις, ε, τα φωτοβολταϊκά θεωρούνται ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, και όλο και περισσότερο ε, χρησιμοποιούνται δασικές εκτάσεις για τη χρήση τους. Στην Γερμανία αποψηλώθηκε δάσος 800 ετών και συχνά βλέπουμε να ε, σκοτώνονται στις ε, ανεμογεννήτριες ε, πουλιά από ήδη σε εξαφάνιση. και ακόμα και νυχτερίδες ή έντομα τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε σκοτώνονται. Επίσης συχνά έχουμε χημικά μείγματα που περιέχουν κάδμιο ή μόλιβδο και γι' αυτό είναι πολύ δηλητηριώδη. Αυτά θέλετε να συνεχίσετε να προωθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρόλα αυτά μιλάμε για προστασία του περιβάλλοντος. Ε, ε, θυσιάζεται η περιβαλλοντική πολιτική. Στα αγγλικά ε, λέμε, έχουμε μια παροιμία που λέει λίγο πολύ ότι δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Πώς το βλέπετε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Thank you very much. I think, uh, Ο κύριος ε, Βόντρα, σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά το θέμα της βιοπικιλότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και Στις προηγούμενες ε, συζητήσεις δεν ήταν πολύ σαφές το αποτέλεσμα, ωστόσο το βασικό πρόβλημα δεν είναι η Ευρώπη. Έχουμε σημαντικές προκλήσεις από χώρες όπως η Κίνα που γίνονται όλο και πιο πλούσιες ε, και Εκεί βλέπουμε διάβρωση των ε, βιοτόπων όπου ζουν ε, ελέφαντες ή τίγρεις. Και θα ήθελα να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι τα στρατηγικά σας σχέδια για τις χώρες όπου η αυξανόμενη ζήτηση ε, ευλάπτει την βιοπικιλότητα. Θα συμβουλεύσουμε τους Κινέζους να μην τρώνε βοηδή και κατόπιν θα τους προσεγγίσουμε με θέματα βιοπικιλότητας ε, ή ε, το εμπόριο του ε, ελεφαντοστούν. Νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να πετύχουμε τα μέγιστα, τελικά δεν θα πετύχουμε τίποτα. Τι μοχλούς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε απέναντι στις χώρες αυτές για να ακολουθήσουν τη Συμφωνία ΣΑΙΤΙΣ και άλλα εργαλεία για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε Βέλλα, κύριε Κομίσιονερ, ε, μιλώντας για την ε, βιοπικιλότητα, ε, και την ε, μαζική εξαφάνιση των ειδών τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Είναι βέβαιο ότι αυτή, αυτού του είδους η ταχύτητα της εξαφάνισης θα οδηγήσει και στην ε, ανθρώπινη εξαφάνιση. η βιοπικιλότητα είναι μια πανανθρώπινη και οικουμενική περιουσία και γι' αυτό τον λόγο είναι ορθή η προσέγγισή σας για την ολιστική αντιμετώπιση με μέτρα από όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Ε, είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην COP15 ε, στην ε, Κίνα θα εξακολουθήσει να ασκεί την πρωτοπορία που οφείλει να ασκεί και στα θέματα αντιμετώπισης της μαλικής κρίσης αλλά και στην, στην βιοπικιλότητα. Όμω θα πρέπει να φροντίσουμε και στα κράτη-μέλη να εφαρμόζονται κοινωτικέ οδηγίες. Η χώρα μου, η Ελλάδα, που έχει το προνόμιο να έχει την μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ε, βρίσκεται στα δικαστήρια με την Επιτροπή σχετικά με την ε, υπερδεκαετή καθυστέρηση να θεσπίσει τους αναγκαίους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διαχείρισης για τους τόπους Natura 2000. Η ριζοσπαστική πρόοδος που επιτεύθηκε στην πολύπλευρη παγκόσμια διπλωματία το 2015, το Παρίσι, η Νέα Υόρκη και το Κίτο, ίσως οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών σε αυτή. Ίσως όμως είναι και αυτή και η αχίλιος πτέρνα τους. Θα πρέπει να δούμε αυτές τις συμφωνίες και να τις στηρίξουμε με πιο δεσμευτικές συμφωνίες, όπως οι εμπορικές συμφωνίες και ειδικότερα τώρα στην Μερκοσούρ θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πέρσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγαμε ε, περίπου 450 εκατομμύρια, ε, δισεκατομμύρια ευρώ βοδινού κρέατος και 821 δισεκατομμύρια ε, σόγιας που αποτελούν και τους μεγαλύτερους, ε, μεγαλύτερες απειλές για τον Αμαζόνιο είτε ως πνεύμονα είτε ως δεξαμενή βιοποικιλότητας. Οπότε κυρίως αυτό θέλω να ρωτήσω την χρήση των δεσμευτικών trade agreements. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Η Άγνες τόνισε τη σημασία του θέματος των ελεφάντων. Θα ήθελα να την διαβεβαιώσω ότι καταπολεμούμε συνεχώς ε, το παράνομο κυνήγι άγριων ζώων ε, καθώς και την παράνομη αποψήλωση και ειδικά όσον αφορά τους ελέφαντες υπήρχε ένα θέμα την προηγούμενη εβδομάδα στην site την ευρωπαϊκή θέση την καθόρισε το Συμβούλιο με απόφαση του Συμβουλίου που ελήφθη με συνένεση. Δεν πληρούν όλοι οι ελέφαντες τις προϋποθέσεις για να μεταφερθούν από το παράρτημα 2 στο παράρτημα 1, όπως συζητήθηκε. Τι επιπλέον μέτρα θέλουμε να λάβουμε. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή νομοθεσία και τα επιπλέον μέτρα που θα πρέπει να λάβουμε αφορούν την εφαρμογή. Πάντα λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επικεφαλής στα θέματα αυτά και η ερώτησή μου είναι εξή: Επικεφαλής πώς όσον αφορά την νομοθεσία ή και όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Και αυτό είναι το βασικότερο ερώτημα. Όταν λοιπόν κάποιος με ρωτάει τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε, θεωρώ ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε ακόμη περισσότερη νομοθεσία, διότι έχουμε καλή νομοθεσία, θα πρέπει να επιδιώξουμε την ε, καλύτερη εφαρμογή. Όσον αφορά την ε, στρατηγική για μη τοξικό περιβάλλον, ε, η προθεσμία μας είναι το 2020. Είπατε ότι η επιστήμη είναι σαφής, συμφωνώ, αλλά... Συχνά οι ανησυχίες μου ξεπερνούν τα όρια της επιστήμης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάντα δίνω το ε, επιχείρημα της ε, μεγάλης ε, κοραλιογενούς ατόλης στην Αυστραλία. Ρωτήθηκαν οι επιστήμονες αν θα αντέξει στην αλλαγή του κλίματος. Πέντε χρόνια αργότερα ερωτήθηκαν το ίδιο πράγμα και απάντησαν ότι όχι, δεν θα μπορέσει να αντέξει. και μέχρι το 2025 θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον αντίκτυπο. Πέρσι ανακοινώθηκε ότι πάνω από το μισό της ατόλης αυτής ε, ήδη έχει νεκρωθεί. Προσπαθώ λοιπόν ε, να σας πω ότι ε, οι εξελίξεις είναι ακόμα πιο γρήγορες από αυτό που μας λένε οι επιστήμονες. Είναι λοιπόν σαφής η επιστήμη, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ακόμη πιο προσεκτική προσέγγιση. Όσον αφορά τα φάρμακα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας και αυτό πάντα μιλώ για την καλή γεωργική πρακτική και τις κακές γεωργικές πρακτικές. Ε, πάντα είμαι σαφής στο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιδοτούμε επιζήμιες γεωργικές πρακτικές και να μην ε, αμείβουμε τις καλές ε, γεωργικές πρακτικές. Δεν κατηγορώ τους ε, γεωργούς, συνομιλώ με τους γεωργούς, θέλω οι γεωργοί να αποτελέσουν μέρος της λύσης, διότι δεν μπορούμε να έχουμε καλή και αποτελεσματική κοινή γεωργική πολιτική χωρίς την ενεργό συμμετοχή των γεωργών. Όταν μιλάμε για φυτοφάρμακα, ε, για λιπάσματα, δεν μπορώ να κατηγορήσω τους γεωργούς, ε, δεν εφήβραν αυτοί τις χημικές αυτές ουσίες, ε, πάλι οι επιστήμονες τις εφήβρανε. Όσον αφορά τα μικροπλαστικά, ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά. Πρέπει όμως να φροντίσουμε οι πολιτικές μας που θα επηρεάσουν όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το μεγαλύτερο μέρος των περιβαλλοντικών πολιτικών μας ε, αντιγράφονται από άλλους σε διεθνές επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλά δεδομένα στη διάθεσή μας ε, προτού λάβουμε αποφάσεις. Ε, στον κύριο Τόρβαλς να απαντήσω, ε, αναφέρατε τον Αμαζόνιο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. Εάν μας ανησυχεί η καταστροφή των δασών και οι πυρκαγιές των δασών, θα πρέπει να μας ανησυχούν παντού όπου και να συμβαίνουν αλλά ναι, όσον αφορά τον Αμαζόνιο, ε, ξεφεύγει από τον έλεγχο η κατάσταση και χρειαζόμαστε ε, πολιτική δέσμευση. Στο Σάρμαλ Σέικ πέρσι, που συζητήθηκε μια παγκόσμια ε, στρατηγική ε, αναζητήσαμε τρία πράγματα. Πρώτον, στόχους, στόχους μετρήσιμους Δεύτερον, χρειάζεται να σταματήσουμε να μιλάμε και να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Χρειαζόμαστε δράσεις. Και τρίτον, χρειαζόμαστε πολιτική δέσμευση υψηλού επίπεδου. Πολιτική δέσμευση από προέδρους και πρωθυπουργούς χωρών. Όταν ε, συναντιόμαστε με τους υπουργούς ε, περιβάλλοντος ε, είναι απολύτως φιλόδοξοι, έχουν όλη την απαραίτητη φιλοδοξία. Όταν όμως επιστρέφουν στα κράτη-μέλη τους, τότε συναντούν προβλήματα με τον Υπουργό Γεωργίας, με τον Υπουργό Οικονομικών, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε πολιτική δέσμευση. Δυστυχώς στη Βραζιλία αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Δεν έχουμε πολιτική δέσμευση υψηλού επίπεδου όσον αφορά αυτές τις πυρκαγιές στα δάση. Στη Μαρή Τουσόν να πω ότι ναι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να προστατεύσουμε τα δάση, όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά παντού. Η Σίλβια ε, ρώτησε εάν ε, συμφωνώ με τη χρήση φινικέλεου και βιοκαυσίμων. Όχι, δεν συμφωνώ. Η λύση που προτείνω εγώ για το μέλλον είναι η ηλεκτρική κινητικότητα, αλλά και πάλι βέβαια θα πρέπει να φροντίσουμε να μην εγκρεμίζουμε δύο εκκλησίες για να χτίσουμε μία, όπως λέμε. Και όσον αφορά το θέμα της ενέργειας, ασκώ πιέσει για να έχουμε παραγωγή ενέργειας όχι μόνο στη γη. Συνήθως ε, μιλάμε για την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια. Ξεχνάμε τι μπορεί να μας προσφέρουν οι ωκεανοί. Εγώ λοιπόν ε, θέλω να προωθήσω την ε, ενέργεια από τον ωκεανό, από την παλήρια, από τα ρεύματα, από τα κύματα του ωκεανού. Μπορεί στην Ευρώπη να έχουμε αρκετές εξελίξεις στο θέμα αυτό, αλλά κάτω από το ραντάρ μπορεί να μην φτάνουν στο φω τη δημοσιότητα. Είναι όμως θέματα ε, τα οποία ε, προωθώ. Ο Αλεξάνδρ ανέφερε την Κίνα. Εγώ τώρα θα μιλήσω ε, ως Καρμεν Βέλα, όχι ως Επίτροπος. Δεν επιτρέπεται να υποτιμάμε το τι κάνει η Κίνα όσον αφορά το περιβάλλον, την άγρια ζωή ασκούμε πιέσεις και έχουμε θετική ανταπόκριση. Ε, είναι τέλειοι σε όλα. Όχι, είμαστε εμείς στην Ευρώπη, δεν νομίζω. Όσον αφορά την Κίνα, πρέπει να σας πω ότι αύριο και την Παρασκευή θα μας επισκεφτεί μια μεγάλη κινέζικη αντιπροσωπεία. Η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα με την οποία καταφέραμε να συνάψουμε συμφωνία εταιρικής σχέσης για τους ωκεανούς. Συμφωνήσαμε δηλαδή να μην ε, συνεχίζουμε τη συζήτηση, αλλά να ενεργήσουμε από κοινού. Να βοηθάμε ένα τον άλλον. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε δεδομένα ε, εικόνες από δορυφόρο και Συνδυάζουμε τα δικά μας στοιχεία με τα δικά τους ε, για τους ε, ωκεανούς ε, και βλέπουμε πώς επηρεάζουν οι ωκεανοί άλλα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε δεν είναι να κατηγορούμε άλλες χώρες. Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε με την κάθε χώρα και να συζητήσουμε ποιος θα είναι ο, ο κατάλληλος και βιώσιμος τρόπος να προχωρήσουμε. Δεν λειτουργεί πάντα, αλλά συχνά λειτουργεί. Όσον αφορά την βιοπικιλότητα, δεν νομίζω ότι... Κάποια χώρα από μόνη της θα μπορέσει να λύσει το θέμα της βιοπικιλότητας. Είναι παγκόσμιο το θέμα. Θα πρέπει όμως να βρούμε και τοπικές λύσεις. Κάθε λύση μετράει. Είχα συναντήσεις με τους Κινέζους και σχετικά με την προετοιμασία της κόπο που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, αλλά θέλαμε κυρίως δράση και δέσμευση σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο από μία-δύο χώρες που να συνάπτουν μεταξύ τους διμερείς συμφωνίες. Νομίζω ότι αναφέρθηκαν ήδη πολλά. Ο Πέτρος ανέφερε ότι ε, αναλάβαμε δράση και όσον αφορά τις περιοχές ε, Natura 2000. Το πρόβλημα με τις περιοχές Natura 2000 δεν ήταν μόνο να εντοπίσουμε, να καθορίσουμε τις ε, περιοχές αυτές. Είχα ρωτήσει αρχικά ποια είναι η συνολική έκταση των περιοχών Natura 2000. Μου είπαν είναι πολύ καλό το ποσοστό, το 20% της Ευρώπης. Και ρώτησα ε, πόσο μεγάλο μέρος αυτών διαχειριζόμαστε σωστά. Περίπου το μισό. Ε, αλλά έτσι δεν προχωράμε και γι' αυτό... Ασκήσαμε πίεση και καταφέραμε από το 50% να φτάσουμε σε 75% αποτελεσματικής διαχείρισης. Προσπαθούμε με αυτοπεποίθηση να προχωράμε. Ε, όμω ε, όμως δεν λειτουργεί αυτή η προσέγγιση, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σύστημα κυρώσεων. Πρέπει να προχωρήσουμε τώρα στον δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ε, κύριε Επίτροπε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Δεύτερος και τελευταίος γύρος ερωτήσεων. Θα ξεκινήσουμε από το ΕΛΚ και την Περνή Λεβάης. Και να σας θυμίσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, ένα λεπτό αναερώτηση έχετε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό δηλαδή συνολικά, μάλιστα. Α, ναι. Καλά, θα τα πω στα πεταχτά. Δεν νομίζω ότι διέφυγε κανένας κατάσταση στους, ε, στον Αμαζόνιο που καλύπτει 30% των δασών σε όλο τον κόσμο και 80% της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένω, έχουμε να κάνουμε μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει τη εποχή όσον αφορά την προστασία της βιοπικιλότητα. Και εσεί, κύριε Επίτροπε, το είπατε. Η βιοπικιλότητα είναι κρίσιμο κομμάτι της ε, κοινή κληρονομιάς των πολιτών. Άρα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην εξαφανιστούν και άλλα είδη. Και τώρα, που λίγει ο χρόνος, θα πω τα εξής. Αυτή η συζήτηση για τις φωτιές, ε, της πυρκαγιάς του Μαζόνιο, βοήθησε την Επιτροπή στην εισαγωγή νέων μέτρων για μια νέα στρατηγική που αναφέρατε και νωρίτερα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, Θεωρούμε πω χρειάζεται κατεπηγόντως να αναλυφθεί δράση. Πώ ε, θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εισαγωγή μέτρων που, θα, που δεν θα πρέπει οικονομικά τουλάχιστον να πλήξουν τις τρίτες χώρες. Μέτρα που είναι αντιπαραγωγικά πρέπει να αποφεύγονται Όπω επί παραδείγματι η αναγκαιότητα για την εισαγωγή τη εμπορική συμφωνία με τι χώρε Μερκοσούρ που πολλοί έχουν αμφισβητήσει. Πρόκειται για μια εσφαλμένη προσέγγιση σε αυτό τη γνώμη σας και στο συγγνώμη ε, γιατί δεν έχω συνηθίσει αυτή την αντίστροφη μέτρηση. Ο Πρόεδρος, σας παρακαλώ να είστε αυστηροί με το χρόνο του ενός λεπτού, γιατί θα προλάβουν και άλλοι, κυρία, ο κύριος Λουένα. Στα γρήγορα να σας πω λοιπόν κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για το πόσο σαφείς είσαστε και να σας πω πως εμείς είμαστε ένα είδος επιθετικό και στο τέλος αυτοκτονικό έτσι όπως δρούμε στον πλανήτη μας. Εκεί θα πάμε. Η Διεθνή Συμφωνία σας παρακαλώ να δώσετε τη μάχη, να είναι δεσμευτική. Η Συμφωνία στην Κίνα πρέπει να είναι δεσμευτική. Για την ΚΑΠ είπατε ε, ναι, υψηλές απαιτήσει, τώρα η γεωργία είτε θα είναι βιώσιμη είτε θα εξαφανιστεί. Για τι πυρκαγιέ, όχι μόνο στην Αμαζονία, χρειαζόμαστε ε, κάτι αντίστοιχο με ό,τι έχουμε σε άλλους ε, κλάδους και για το Μερκοσούρ. Ο Μπολσονάρο θα συμμορφωθεί. Και τέλος, έχουμε... Με, έχουμε αυτή τη στιγμή μία επιδημία στα πουρνάρια στην Ισπανία που μπορεί να τα εξαλείψει, οπότε θα ήθελα να μου πείτε για τα είδη κουέρκους, αν έχετε σκοπό να πάρετε κάποια μέτρα. Thank you. For renew, Nicolas Stefan. Nicolas. Παρακαλώ. Κύριε Βέλα, φαίνεται πως ε, Υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της ε, πραγματικότητας της προστασίας ε, της βιοποικιλότητας. Έχουμε ε, νομοθεσία μένα, αλλά δείχνουμε διαφορία και καταστρέφουμε την, το, ενδυμα, το πολλών ειδών. Η Ρουμανία, η πατρίδα μου, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό παρθένων δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μεγάλες όμως καταστροφές ενώ υπάρχει νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν φέρνει αποτελέσματα αυτή, δεν είναι ουσιαστική. Έχουμε ένα κόστος ετήσιο από μη, εφαρμογή της νομοθεσίας που ανέρχεται ακόμα και στα 55 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επομένως πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να προστατεύσουμε αυτές τις περιοχές. Πώς μπορούμε να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις δράσεις μας κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, τι είδου μέτρα σκοπεύετε να αναλάβετε εσείς και οι συναδελφοί σας, τι είδου σχέδια έχετε για την διάσκεψη των Εθνών του 2020 για τη βιοπικιλότητα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Πράσινη. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κύριε Βέλα. Ευχαριστώ για τα λόγια σας κύριε Παύλος. Το Ινστιτούτο της Στοκχόλμης ε, για την αντοχή έχει, έχει καταγράψει εννέα όρια βιοπικιλότητας και αυτό που συζητείτε αυτή τη στιγμή είναι η απώλεια βιοπικιλότητας με την επιτάχυνση κατά 100 και 1000 φορές της εξαφάνισης ειδών. Η εξαφάνιση ειδών είναι κάτι το απολύτως οριστικό πάνω στον πλανήτη Γη. Δεν μπορούμε να προστατεύουμε λοιπόν ε, ακόμα και μικρά κομμάτια γης, φυσικά πάρκα και οι περιοχές Natura 2000 με αποσπασματικά μέτρα. Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση με τη γεωργία, με τις πόλεις, με την προστασία των υδατινών πόρων, ε, με τις μεταφορές του χρόνου στην Κίνα, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ζητήσει ένα δεσμευτικό πλαίσιο για να προστατεύσουμε ε, τη φύση και να εξασφαλίσουμε τους στόχους μας πριν ολοκληρωθεί ο ερμαγεδόν αυτός. Θα υπάρχουν σαφείς ε, γραμμές για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει μια διεθνή συμφωνία. Η βιοπικιλότητα εξασφαλίζει το απαραίτητο ελάχιστο για την επιβίωσή μας. Ας μην το καταστρέψουμε. Έχουμε ακόμα καμιά εδώ ερωτήσεις για την στρατηγική για το 2020 και για το ποια θα είναι η θέση σας στην ΚΟΠ στην Κίνα. Οπότε καλό θα ήταν αυτό να τα βάλετε, ε, να τα ομαδοποιήσετε στην απάντησή σας. ID, Σίλβια Λίμερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήξερα ότι είχε έρθει και πάλι η σειρά μου. Ε, σας αξιοποιήσω λοιπόν την ευκαιρία να σας κάνω για άλλη μια φορά την ερώτηση. Είχατε αναφερθεί στην ε, αύξηση των, ε, στην χρήση νέων πόρων καυσίμων. Μιλήσατε για την χρήση των ε, υδάτων των ωκεανών. Είναι δυνατόν αυτό να συνδυαστεί με την προστασία της φύσης και κάτι ακόμη στο οποίο δεν απαντήσατε. Η χρήση των φωτοβολταϊκών που διαδίδεται όλο και περισσότερο δεν οδηγεί σε εξαφάνιση ειδών. Και μήπω τελικά αυτό σημαίνει και το τέλο μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. ECR, παρακαλώ. Ζαλεύσκα. Κομισάζου. κυρία Ζαλεύσκα. Κύριε Επίτροπε, με βλέπετε? Μιλήσατε εσείς για το ότι δεν έχουμε πετύχει τους στόχους για την βιοπικιλότητα και πρέπει εδώ να σας απευθύνω μια σειρά από ερωτήσεις. Είναι σημαντικό, καταρχήν, να μου πείτε ποιες ήταν οι επιπτώσεις γιατί μας υπενθυμίσατε πως αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε όλα αυτά για την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης δεν θα έπρεπε να διαπιστώσουμε τι γίνεται με τα κονδύλια που θα πάνε για να στηρίξουν τη βιοπικιλότητα, πώς θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, η πρωτοβουλία η οποία ε, <laughs> ονομάζεται Συμφωνία των Καρπαθίων Τσεχία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σερβία, Ουκρανία και Πολωνία, που είναι η δική μου χώρα, προσφέρει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πρόπτικες. Okay, so Mick uh, for the e. e? κύριος είπατε στα εισαγωγικά σας uh, σχόλια πως ξεπεράσαμε για τις ε, υποπροστασίες θαλάσσιες περιοχές ε, τα όσα θα έπρεπε να έχουμε κάνει. Όμως, ποια είναι η έκταση αυτών των θαλασσών και τι ποσοστό της συνολικής θαλάσσιας έκτασης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι. Και πώς γίνεται η διαχείριση αυτών, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για την βιοποικιλότητα. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, έχει μια διεθνή υποχρέωση να ορίσει 10% της θάλασσάς της ως προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Αλλά μετά από μια μελέτη που έκανε το Wildlife Trust στην Ιρλανδία, μόνο το 3% αυτής της τεράστιας θαλάσσιας περιοχής προστατεύεται με ειδικό τρόπο. Και είμαστε οι δεύτεροι από το τέλος για τα κράτη-μέλη ε, στη δημιουργία ε, προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών. Πιστεύετε πως η Ιρλανδία δεν κάνει ότι θα έπρεπε. Συμφωνείτε πως αυτό το 10% στόχος θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα πάνω εν ώψη της ε, παγκόσμιας έκθεσης αξιολόγησης της και του γεγονότος πως χειροτερεύει με ε, ιστορικό τρόπο η βιοπικιλότητα σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ. Έλκα. Κύριε Επίτροπε, στις 29 Ιουλίου μιλήσαμε στην ανοιχτή ημέρα για τα όσα γίνονται κάθε χρόνο σε επίπεδα κατανάλωσης πλανητικών ε, πόρων. Κάθε χρόνο τρώμε 1,75 πλανήτες γη. Κάθε χρόνο αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Κάθε μέρα μειώνονται, κάθε χρόνο μειώνονται οι βροχοπτώσεις στο νότο της Ευρώπης. Ερημοποίηση. Έλλειψη βιοπικιλότητας. Η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος, η Ισπανία. Είναι από τις χώρες που επηρεάζονται πιο πολύ από την ερημοποίηση και κινδυνεύει ακόμα πιο πολύ η βιοπικιλότητα μας. Πάνω από το 50% της πορτογαλικής επικράτειας κινδυνεύει και η ερημοποίηση είναι για μας η μεγαλύτερη απειλή για την βιοπικιλότητα. Τι χρειάζεται λοιπόν, πολιτική συστράτευση και υποχρεωτικές ε, ρήτρε για να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Επίτροπο εκπροσωπώντα του σοσιαλιστές και να σα πω το εξή. Έχουμε το άρθρο 349 τη συνθήκη και λαμβάνοντα υπόψη τη στενή σχέση που έχουν οι, ε, οι νησιωτικές περιφέρειες της Ευρώπης ε, και οι απομακρυσμένες περιοχέ με τη θάλασσα, τι θα κάνετε για να διατηρήσουμε εν ζωή τα θαλάσσια είδη. Υπάρχουν οικονομικά και κοινωνικά θέματα που συνδέονται με το θαλάσσιο κλάδο σε αυτές τις απομακρυσμένες περιοχές. Δεύτερον, κλιματική αλλαγή έχουν εισαχθεί νέα είδη σε συγκεκριμένες περιοχές. Κάτι το οποίο έχει διαταράξει τη βιοποικιλότητα στις περιοχές αυτές, ε, γιατί τα αυτόχθονα είδη ε, κινδυνεύουν. Έχετε εποπτικό μηχανισμό για να ελέγξουμε αυτές τις, ε, αυτά τα είδη, τα οποία ενδεχομένω είναι και ξενιστές ασθενειών. Πώς θα προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους. Caroline Renew. Caroline, Renew. Ευχαριστώ πολύ. Η αξιολόγηση φέτος για τη βιοπικιλότητα μας, απειλεί, μας ενημερώνει πως μας απειλεί μία χωρίς προηγούμενο μείωση της βιοπικιλότητας σε όλο τον πλανήτη και τα τελευταία νέα έχουν να κάνουν με τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, αλλά έχουμε θέμα και με τις θάλασσες. Η βιοπικιλότητα στους ωκεανούς μας είναι κομβική σημασία για όλους μας. Κάθε μέρα 60.000 εμπορικά τάνκερ ε, πλέον στους ωκεανούς μας. 60.000 σκάφη ε, που εκπέμπουν ήχους, ε, που θανατώνουν ε, ασπόνδυλα ή θηλαστικά. Και με τον τρόπο αυτό εμείς ε, καταστρέφουμε τα υποθαλάσσια οικοσυστήματα. Τεχνική για να μειωθεί αυτή η χορύπανση υπάρχει. Έχουμε τη βούληση, για παράδειγμα, ένα 10% μείωση της ταχύτητας των σκαφών μπορεί να μειώσει την χορύπανση κατά 80% ή την εκπομπή ήχων. Τι θα κάνετε εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μειωθεί η χορύπανση από τα πλοία. Πώς θα πιέσετε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση, πώς θα τα υποχρεώσετε να λογοδοτήσουν για να διατηρήσουμε την πολύτιμη βιοπικιλότητα ποιότητα των ωκεανών μας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κάνευ από το ΕΛΚ. Thank you. Uh, for 12 years of European membership... Ο κύριος Κάνευ. Η βουλγαρική κυβέρνηση τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μέλη έχει εφαρμόσει μόνο 12 από τις 200 αποφάσεις για τα ενδιαιτήματα Habitat natura, ε, με συγχωρείτε. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια και στους μικροκτηματίες και στους μεγαλοκτηματίες και στους επενδυτές. Δεν ξέρουν τι θα γίνει με την οδηγία για τα ενδιατήματα και ενώ υπάρχουν κανόνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε αυτά αποτελέσματα. Έχουμε πάρα πολλές οριζόντιες αναφορές και καταγγελίες για αυτές τις παραβιάσεις. Χρόνια περιμένω να λάβουν μια απάντηση και μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Κάποια έφτασαν το 2009 στα αυτιά της Κομισιόν. Άρα λοιπόν, και αυτή είναι η βασική μου ερώτηση, προφανώς έχουμε προβλήματα επιβολής εδώ στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, Θέλω να σας πω πως βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντική βιοποικιλότητα στη Βουλγαρία και έχουμε πολλές προσδοκίες πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δράσει αποφασιστικά έτσι ώστε ε, να τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά σπάνια αυτές οι προσδοκίες γίνονται πραγματικότητα. και δημοκράτε, Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Βέλα και να ρωτήσω για άλλη μια φορά την, ιστορία, την ερώτηση σχετική με το grooming. Είχαμε λοιπόν ε, στην υπόθεση αυτή του, της Συμφωνίας των Παρισίων να ε, προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική περιγραφή του όρου για να φέρει τα αποτελέσματα η Συμφωνία των Παρισίων που περιμένει ο κόσμος και που έχουμε διεκδικήσει κι εμείς. Πρέπει να έχουμε ουσιαστικούς στόχους και γι' αυτό ερωτώ. Ένα κομμάτι σημαντικό πιστεύω της ε, αρρώσιμης γης αλλά και των παράκτων περιοχών πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για εκμετάλλευση, δεν πρέπει να προστατεύεται η φύση και οι πληθυσμοί η εξαφάνιση ειδών πώς μπορεί να αποτραπεί η Επιτροπή, κύριε Βέλα, πώς μπορεί να παρέμβει και τι είδους στόχους να προσδιορίσει. Και αν έχει πράξει κάτι τέτοιο, τι αντιδράσει έχει δει μέχρι τώρα εν ώψη μιας νέας συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Σύνσήτηση από τους μη εγγεγραμμένους, τελευταία ερώτηση. Επίτροπε, μιλήσατε για την προστασία των δασών του Αμαζονίου, που είναι τόσο απαραίτητη, διότι τι χρειαζόμαστε, τα χρειαζόμαστε τα δάση αυτά για να επιβιώσουμε ως ανθρωπίνο είδος. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να γίνουν πυρκαγιά στην Αμαζόνιο για να δούμε τι μεγάλε καταστροφέ. Μέσα σε 10 χρόνια στην Κροατία έχουν χαθεί δεκάδε χιλιάδε εκταρίων με αποψήλωση ακόμα και σε περιοχές προστατευόμενων δασών, λόγω της διαφθοράς, λόγω του ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση ούτε καν στην Κροατία να προστατέψει τα δάση. Πώς μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε να τα προστατεύσουμε τα δάση του Αμαζονίου, που απέχουν και δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, ε, όταν δεν μπορούμε τα δικά μας δάση να προστατέψουμε. Ο πρόεδρος πολλές ερωτήσεις για τον Αμαζόνιο, για την αποψήλωση, για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω μόνο ότι για αύριο προβλέπουμε ένα ειδικό κομμάτι στη συζήτησή μας, στη συνεδρίασή μας για τα θέματα αυτά. Ελπίζω να σας ξαναδούμε βέβαια ε, αγαπητοί συνάδελφοι, να διατυπώνετε τις ίδιες ερωτήσεις, ώστε να εγγραφούν ε, στις απαντήσεις που θα δώσει η Επιτροπή εν ώψη του ανακοινοθέντος της. Και γι' αυτό, κύριε Βέλα, εάν θέλετε, επικεντρωθείτε περισσότερο σε άλλα θέματα και όχι στην αποψήλωση, που όπως είπα αύριο θα μας απασχολήσουν ούτως ή άλλως. Και για την COP15 ε, του 2020 θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Έχει γεννήσει πολλές προσδοκίες. Παρακαλώ. Ναι, Ας ξεκινήσω από την COP15. Καταρχάς, όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία του να έχουμε ένα πλαίσιο βιοπικιλότητας για μετά το 2020 και θέλουμε όχι απλά ένα νομοθετικό πλαίσιο, θέλουμε ένα σχέδιο δράσης. Η βιοπικιλότητα είναι σημαντική όχι μόνο για την ε, Συμφωνία του Παρισιού ή για τους στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι σημαντική και σε εκείνο το πλαίσιο, αλλά είναι σημαντική και ε, ως αυτός σκοπός. Όλοι δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα. Συνεχίζεται όμως η απώλειά της με μεγάλες ταχύτητες και γι' αυτό χρειάζεται παγκόσμια δράση. Έχουμε ξεφύγει από την ασφαλή περιοχή που ήμασταν και θέλουμε ε, η COP15 να φτάσει στο επίπεδο του Παρισιού. Από την Σύμβαση Βιοπικιλότητας 15 ε, θέλουμε στόχους ε, με προθεσμίες, στόχους μετρήσιμους και να καταφέρουμε να αναχαιτήσουμε την απώλεια βιοπικιλότητα ε, με έναν στόχο παρόμοιο με τον ε, στόχο των δύο βαθμών Κελσίου ε, στο κλίμα. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε δράση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι. Αυτό κάνουμε στι διασκέψεις για τους ωκεανούς. Ε, δεν συζητάμε απλά, ο καθένας πρέπει να υποβάλει στόχους και κατόπιν έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης που εξετάζει εάν έχουν ε, ε, πραγματοποιηθεί η δεσμεύσει και έχουμε πολιτική δέσμευση υψηλού επίπεδου και γι' αυτό έχουμε πάει στα Ηνωμένα Έθνη το θέμα της βιοποικιλότητας με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε και για τους ωκεανούς. Και χρειάζεται να ακούμε τη φύση, να μην περιμένουμε απλά καινούριε εκθέσει. Κάθε φορά που συζητάμε κάτι, ακούμε ότι α, εντάξει, περιμένουμε μια έκθεση σε τρία χρόνια, α την περιμένουμε. Καλέ οι εκθέσει, αλλά απλά επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη μα λέει η φύση. Είχαμε την ε, έκθεση για την κατάσταση της φύσης, ε, την έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Είχαμε την ενδιάμεση έκθεση που συνδέεται με τις ε, οδηγίες για τη φύση. Δεν νομίζω όμως ότι θα πρέπει να προσέχουμε πιο πολύ τις εκθέσεις και να ξεχνάμε τη φύση. Το άλλο στο Σάρμελ Σέικ ήταν ότι όλοι μπερδεύονται όταν τίθενται ερωτήσεις του τύπου τι σκοπεύετε να κάνετε. Αν ρωτήσετε κάποιον τι σκοπεύεις να κάνεις, αμέσως επικρατεί σύγχυση. Γιατί? Γιατί να επικεντρωθούμε στο τι πρέπει να κάνουμε και να μην επικεντρωθούμε στο τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όλες αυτές οι περιβαλλοντικές εκθέσεις μας δείχνουν τις βασικές αιτίες της απώλειας βιοπικιλότητας, αλλαγή χρήση της γης, ε, γεωργία. Εάν γνωρίζουμε ποιες είναι οι αιτίες, εάν γνωρίζουμε τι προκαλεί την ε, απώλεια βιοπικιλότητας, ε, τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτούμαστε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο το τι πρέπει να κάνουμε. Είμαι αισιόδοξο όσον αφορά το μέλλον. Να σας αναφέρω κάποιες από τις δράσεις της Ευρώπης για την αναχέτηση της ε, απώλειας βιοπικιλότητας. Ε, καταρχάς, θέτουμε το θέμα αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα από τα προβλήματα που είχαμε και δεν καταφέραμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε μέχρι το 2010 και το 2020 αντίστοιχα, ε, το πρόβλημα ήταν ότι η διεθνής κοινότητα δεν νομίζω ότι γνώριζε αρκετά το πρόβλημα. Τώρα που υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση είμαι πιο αισιόδοξο ότι θα επιτευθούν οι στόχοι που θα τεθούν. Αναφέρθηκα στο σχέδιο δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία. Είχαμε την πρωτοβουλία για τους επικονιαστές για να ε, αναχαιτήσουμε την εξαφάνιση των επικονιαστών και έχουμε ε, έγγραφα προσανατολισμού ώστε να έχουμε ε, τις ε, κατάλληλες υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Σάρα νομίζω ανέφερε τον κατάλογο των χωροκατακτητικών ειδών, έναν κατάλογο τον οποίο επικαιροποιούμε συνέχεια επιδιώκουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, διότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και στην εξέβρεση άλλων λύσεων. Ε, θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις λύσεις που βασίζονται στη φύση, δεν χρειάζεται να ε, εφεύρουμε νέα πράγματα. Έχουμε επίσης ε, μια διευκόλυνση για την χρηματοδότηση προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τη φύση και επίσης ε, έχουμε ένα πρόγραμμα για την βιώσιμη χρηματοδότηση ώστε να φροντίσουμε κάθε πρόγραμμα να προστατεύει και όχι να καταστρέφει τη βιοπικιλότητα. Επίσης είμαστε πολύ δραστήριοι όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου ε, κυνηγιού ε, άγριων ζώων, της παράνομης υλοτομίας και της ε, παράνομης ε, και αναρχής ε, και μη ρυθμισμένης αλληλείας. Είχε υποθεί ότι θα μειωθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος σε αλλά αυτό το αποφύγαμε και επίσης έχουμε και τον ρόλο των κρατών μελών. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς τα πάντα από την Ένωση και να μην περιμένει τίποτα από τα κράτη-μέλη. Έχουν λοιπόν και τα κράτη-μέλη ρόλο να παίξουν και τα στηρίζουμε. Συνεργαζόμαστε μαζί τους ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται με την νομοθεσία μας για τη φύση και επίσης ε, ε, έχουμε θεσπίσει διαλόγους με τα κράτη-μέλη για την φύση και τη βιοπικιλότητα. Και φυσικά όταν υπάρχει ανάγκη επιβολής του νόμου είναι και αυτό ένα θέμα που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Δεν ε, θα αναφερθώ τώρα στις περιοχές Natura 2000, ε, αλλά ακόμα και όταν μιλάμε για τη βιοπικιλότητα, επικεντρωνόμαστε κυρίως στη βιοπικιλότητα στη στεριά, αλλά εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στους ωκεανούς, στα πάντα. Απογοήτευση για μένα στις συζητήσεις του Παρισιού ήταν ότι συζητούσαμε την αλλαγή του κλίματος, ενώ οι ωκεανοί που μας δίνουν το 50% του οξυγόνου μας, απορροφούν το 50% του διοξιδίου του άνθρακα μας, ε, ε, όπου μένει το 50% των ειδών του πλανήτη, δεν αναφέρθηκαν καθόλου. Μιλούσαμε λοιπόν, ε, τώρα λοιπόν που συζητάμε για την βιοπικιλότητα, σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι ε, έχουμε εξίσου ε, πολλή βιοπικιλότητα στους ωκεανούς, την οποία θα πρέπει να σώσουμε όσο έχουμε και στη στεριά. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ πάντως για την συζήτηση και οι συνεργάτες μου θα ε, σας ε, δώσουν τις δικές τους παρουσιάσεις αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πως ε, μιλήσατε όχι μόνο με το μυαλό, αλλά μιλήσατε και με την καρδιά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτό. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή, δύο λεπτά, και μετά θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Kif inti dalli? Kif morna? لا Le من وحياي Please, colleagues, we are going to start the vote. So please, if you could join your seat. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Merci, je vais... I'm going to switch to French, so... Και θα μιλήσω γαλλικά. Γι' αυτό περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας αν χρειάζεται. Έχουμε λοιπόν δύο ψηφοφορίε. Η πρώτη αφορά το Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Δημοσιονομικό έτος 2020 και η δεύτερη τη Δημοσιονομική Διαδικασία 2020. Αρχίζουμε με το Γενικό Προπολογισμό. Γνωμοδότησή μα για το Γενικό Προπολογισμό 2020. Έχετε τα έγγραφα. Πρωτοβολογία πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές και απερίφθη. Δύο. Σε τμήματα. Το πρώτο τμήμα παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Προφορική τροπολογία του εισηγητή δηλαδή εμού του ιδίου, ως προέδρου, υπό την ιδιότητα αυτή, αντί για το to be set at least at 50%, to be set at 40%, αντί για 50%, 40%. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα την προφορική τροπολογία, αν δεν υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Την ψηφίζουμε λοιπόν 40%. Αυτό ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ του 40%. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Και άρα καταπίπτει η αρχική τροπολογία. Άρα το κείμενο υιοθετείται με ένα 40% στη διατύπωση. Υπαριθμόν 3. Υπέρ κατά αποχές το ΕΛΚ δεν βλέπω τη στάση υπέρ μάλιστα εγκρίνεται λοιπόν τέσσερα υπέρ κατά αποχές σε επαληθεύσουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά αρχίζουμε Πέρας. Όχι, όχι. Παραμένει ανοιχτή η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέντε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έξι υπέρ. Κατά. Αποχέ απερίφθη. Παρα, ε, ε τροπολογία υπαριθμών 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 έχει, έχει αποσυρθεί όχι, πρόκειται για διαγραφή 11 την ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 σε τμήματα πάλι πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα της, δεκάτα της τέταρτης τροπολογίας υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ Μια κάρτα που δεν δουλεύει. Έχετε κάποιον άλλον εσείς. Έχετε άλλο συναδελφό σας που μπορεί να αναλάβει να ψηφίσετε στις κυρία Στόγια. Καλώς. Λοιπόν. Μήπως στην άλλη πλευρά, στο άλλο μηχάνημα. Καλά, τότε θα υπολογίσουμε την ψήφο σας. Ε, στα πρακτικά. Με βάση τόσα ψηφίσεις και ομάδα σας. Μέστε. Απεριφθεί. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 έχει καταπέσει ή 18 τώρα υπέρ με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος επιστρέφω στη 17 και εξηγώ ότι έχει καταπέσει επειδή νεκρήθη η 16 και έτσι πάμε στη 18η τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά. Αποχές. Απεριευθεί. 21 υπέρ. Υπέρ. 21 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε την 21. Πέρας. Απερίφθη. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 24. Έχει αποσυρθεί. 25 υπέρ. Κατά. αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε πέρα στις ψηφοφορίες και εγκρίνεται 27 υπέρ κατά Αποχές και επαληθεύουμε. Πέρας. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική, ονομαστική και έτσι ο καθένας ξέρει τι έχει ψηφίσει. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Βλέπω κάποιοι ακόμα να μην έχουν ψηφίσει. Μας λείπει μία ψήφος. Ωραία, ψηφίσατε κι εσείς. Πρόεδρε, παρακαλώ, μπορείτε για τα πρακτικά να καταγράψετε πώς υπερψήφισα. Δεν είναι ότι ξέχασα την κάρτα μου, αλλά πήρα την περσινή. Και δεν δουλεύει. Καλώς. Άρα 60 υπέρ. Και πάμε στη δεύτερη ψηφοφορία για σήμερα. Νομοσονομική διαδικασία 2020. Ακολουθούμε τη σειρά την αριθμητική των τροπολογιών 5400, 5475 κτλ. Στην γνωμοδότηση. κοινέ οι 5400 και 5475 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνονται 5420 υπέρ. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, επανέρχομαι, είναι on block ομού με την 5423. 5420 και 5423 ομού υπέρ. Κατά. Απερίφθη. Σαν. 54, 42 και 54, 04. Όχι χωριστά. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 54, 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54, 04 καταπίπτει αφού εγκρίθηκε η 54-42. Ψηφίζουμε την 54 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 5405 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Την 54-23 την ψηφίσαμε μαζί με την 54-20 πιο πριν, άρα δεν χρειάζεται να την ξαναψηφίσουμε. 54-66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Πέρας. Περίφθη. 54-78 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 54-41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54-46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54-43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54-22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54-64 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται μαζί με την 54-76, την οποία είχαμε εν μπλοκ. Η επόμενη 5439 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 54-40. Εδώ και πάλι έχουμε προφορική τροπολογία που έχει καταθέσει ο κύριος Φερέιρα. Για την προφορική λοιπόν θα ψηφίσουμε εκτός αν υπάρχουν αντιδράσεις. Ποιο είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας αυτής. Κατά. Απορρίπτεται ε, η προφορική της εκδοχή. Περνάμε στην 5445 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5447 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54-56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54-57 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 54-58 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται 54-59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 54-60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 54-48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 5449 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5450 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5451 υπέρ κατά Εδώ θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω πως απερίφθη. Πέραση ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να επαληθεύσω. 54-52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54-36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριπεται 54 54-37 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε και εδώ πέρας εγκρίνεται 54-67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54-25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για δύο ταυτόσμες, την 5409 και την 5426 μαζί υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν μπόρεσα να σας μετρήσω, με συγχωρείτε. 54-65 είναι σε μπλοκ με την 54-77 ε, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 54-10 και 54-27 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54-44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54-62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54-63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54-74 μαζί μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 5412, 54-29... Μπορείτε να μας αφήσετε το χρόνο να ψηφίζουμε. Πηγαίνετε λίγο γρήγορα, παρακαλώ πολύ. Ωραία, λοιπόν, θα το ξαναδούμε. Είμαστε 54-12, 54-29, 54-73. Είναι τρεις ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54-30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54-38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 54-34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54-01 54-19 54-55 ταυτόσιμες ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 54-02 54-21 54-54 υπέρ κατά 54-03 αποχές εγκρίνονται. 5403, 5470 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 5406, 5424, 5469 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. 54-07-54-68 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνονται. 54-08-54-53 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνονται. 54-13-54-31 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνονται. 54-14-54-32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 54-15, 54-33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 54-16, 54-35, 54-71 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 54-17, 54-79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται 54-18, 54-72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Την δύο τελευταίες τις έχουμε ήδη ψηφίσει προηγουμένως α, unblock, οπότε τελική ψηφοφορία που δεν θα γίνει. Α, δεν θα γίνει. Οπότε το ρυθμίσαμε έτσι. Σας ευχαριστώ για την ε, εμπειρία αυτή που ήταν μια πρώτη ε, πειραματική ψηφοφορία. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9.